Good evening. Καλησπέρα σας, κύριε Επίτροπος. Καλώς ορίσατε. Ξεκινάμε την νυχτερινή συνεδρίασή μας. Καλώς ορίζω τον Υπουργό κύριο Χόντρατ. Δεν ξέρω πού εκπροσωπείται καλύτερα το Συμβούλιο, Κομισιών ή το σώμα μας, αλλά μέσα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Έλαβα κάποιες αιτήσει ε, για αλλαγές ε, σε διακοινοβουλευτικές επιτροπέ και σε αντιπροσωπείε Ο κατάλογος ε, των ορισμών θα επισυναυθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως. Εάν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξουν ενστάσεις, αυτοί οι διορισμοί θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένοι.